την εντολή των συναδέλφων Γκράς Βάντερ Χάινς, του κυρίου ε, Στέφανο Μάουλου, του κυρίου Νικολάου Χουντή και του κυρίου Άουκ Ζέλστρα και πρότεινε να εγκριθούν και να κηρυχθούν έγκυρα οι εντολές από τις 9 Ιουλίου, από τις 13 Ιουλίου, από τις 20 Ιουλίου και από την 1η Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Γι' αυτό προτείνω να ε, θεωρήσουμε την έγκυρη εντολές. Δεν ξέρω αν διαφωνεί κανείς σας. Διαπιστώνεται λοιπόν η εγκυρότητα των εντολών. Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές ε,